Καλημέρα κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Αν θέλετε μπορούμε, μπορείτε να καθίσετε πρώτον να αρχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων μετά. απευθύνω το καλώ ορίσατε στον Επίτροπο κ. Ανδρουκάητη. Τον ευχαριστώ για την έλευσή του για να συζητήσουμε τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. Έχει ενδιαφέρον το θέμα αυτό για μας και γνωρίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα μόλις αναθέσαμε την ε, σύνταξη της εκθέσεως ε, στους σοσιαλιστές και δημοκράτες, αν και δεν έχουμε ακόμα το όνομα του εισηγητού ή της εισηγητρίας. Θα το έχουμε όμως σύντομα. Είναι ενδιαφέρον το θέμα και αναμένουμε να αρχίσουμε την εργασία που γνωρίζω ότι είναι σημαντική και για εσάς, δηλαδή να μπορέσει να εγκριθεί ε, η σχετική νομοθεσία πριν από το τέλος της περίοδου. Ας ακούσουμε πρώτα εσάς και μετά θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να θέσουν ερωτήσεις εφόσον το επιθυμούν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που εμφανίζομαι σήμερα ενώπιόν σας για να μπορέσω να παρουσιάσω τη σημαντική αυτή νομοθετική πρόταση που έχει ως στόχο να ενισχύσει την συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Μακρά ήταν η πορεία για να φτάσουμε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα μας ενθαρρύνουν τα θετικά σχόλια που έχουμε ακούσει έως τώρα. Μετά από 20 χρόνια οικειοθελούς συνεργασίας στον χώρο αυτό και εκτεταμένες περιόδους προβληματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει μια, ένα σχέδιο νομοθετικής πρότασης ήδη από την 31η Ιανουαρίου για την συνεργασία για θέματα τεχνολογίας υγείας. Φιλόδοξη πρόταση η οποία θα αποδώσει προστιθέμενη αξία στις ε, χώρες μέλη, βεβαίως και στους ασθενείς και στην βιομηχανία. Η πρόταση θα διευκολύνει ε, περαιτέρω την αντικειμενική αξιολόγηση βασισμένη σε ενδείξεις της ε, τεχνολογίας υγείας. Πρώτα, με τεχνολογίες υγείας ε, εννοούμε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, ιατρικών, ε, ιατρικών συσκευών, διαγνώσεως in vitro και ούτω καθεξής. Θέλω να διευκρινίσω κάτι ωστόσο από την αρχή, διότι αντιλαμβάνομαι ότι καμιά φορά προκαλείται σύγχυση σχετικά με το τι σημαίνει η συντομογραφία HTA. Μιλάμε για την ε, post-marketing φάση των τεχνολογιών υγείας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εν προκειμένου είναι η αξιολόγηση του πώς τα προϊόντα υγείας και οι παρεμβάσεις αποδίδουν, λειτουργούν στην πραγματική ζωή. Η HTA δεν σημαίνει ε, αξιολόγηση μόνο της απόδοσης ενός εργαλείου, ενός μηχανισμού, αλλά και τη θεραπευτική προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με υφιστάμενες θεραπευτικές τεχνολογίες. Διότι οι τεχνολογίες υγείας είναι ένα ισχυρό εργαλείο που θα μας επιτρέψει, το HTA μάλλον, να κάνουμε τη σχετική αξιολόγηση. Εν τέλει δε θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές υγείας να εντοπίσουν πραγματικά καινοτόμες τεχνολογίες και να τις αξιοποιήσουν και να κάνουν και τις σωστές επιλογές υπέρ των ασθενών. Καμιά φορά βλέπει κανείς καινοτομίες που είναι καινοτομίε μόνο στα χαρτιά, όχι όμω στην πραγματική ζωή. Και η HTA θα μα διευκολύνει να αξιολογήσουμε την πραγματική καινοτομία στην πραγματική ζωή και θα φέρει και διαφάνεια και θα διευκολύνει και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμε τεχνολογίε υγεία. Ταυτόχρονα δε θα συμβάλλει στην βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Όπως ε, το περιγράφει και το κοινό δίκτυο δράσεων, η HTA μπορεί να χωριστεί σε δύο τομείς, τον κλινικό τομέα και τον μη κλινικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, σε εννέα υποσημεία, ξεκινώντας δηλαδή από τον κλινικό τομέα, όπως εντοπισμός των προβλημάτων υγείας και της τρέχουσας χρήσης της τεχνολογίας, θέματα ασφαλείας κλπ και βεβαίως και στον μη κλινικό τομέα, όπως οικονομική αξία, κοινωνικές πτυχές, διοντολογικές πτυχές και ούτω καθεξής. Ορισμένα παραδείγματα της τεχνολογίας τα βλέπετε στην παρούσα διαφάνεια, όπου ορισμένα καθίστανται δυνατά και ε, στην βάση του δικτύου κοινών δράσεων που έχει ιδρύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα σημαντικές θεραπείες για ε, τον καρκίνο ή για τα εμβόλια. Αυτά γίνονται τώρα σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο από περισσότερες, περισσότερες από 50 ε, συμβούλια σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε διαφορετικές χώρες μέλη με χρήση διαφορετικών μηχανισμών. Οι χώρες μέλη κάνουν την κλινική αξιολόγηση μετά από την διαδικασία διάθεσης στο εμπόριο στην αγορά. Επομένως, τεχνικές και αξιολογήσεις ιατρικών ε, ε, μηχανισμών γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Γίνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο και 21 χώρες μέλη αξιολογούν συστηματικά τις ιατρικές συσκευές. Εν τέλει βλέπουμε ότι είναι κατακαιρματισμένη η τεχνολογία αξιολόγησης των ε, ιατρικών τεχνολογιών για την ώρα. Αυτό αποβαίνει σε βάρος και των χωρών μελών και των ενδιαφερομένων μερών. Έγινε διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους για να συλλεχθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία και πέραν του 2020 σχετικά με την HTA. Λάβαμε 300, 249 απαντήσεις. 50% από τη βιομηχανία και 25% από άτομα, από πολίτες, οι περισσότεροι από αυτούς, 87% όλων θεωρούν την προοπτική της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την HTA χρήσιμη ή εν πάση περιπτώσει χρήσιμη σε κάποιο βαθμό. Από την έγκριση της προτάσεως χαίρομαι διότι πολλοί, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν θετική την αυτή πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας. Όλες οι δυνατές ε, προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας έχουν ληφθεί υπόψη. Ένας αριθμός μελετών έχουν ανατεθεί για να διασφαλιστεί ότι θα έχουμε τα αναγκαία δεδομένα για να συντάξουμε τη σχετική νομοθετική πρόταση. Παρά τις πολλές επιτυχίες που έχουμε ως τώρα, έχουν διαπιστωθεί ωστόσο και σημαντικές ελλείψεις. Ε, υπάρχει απόκληση τεχνολογιών, διαδικασιών και έλλειψη βιωσιμότητας του τρόπου συνεργασίας που χρησιμοποιείται ως τώρα. Αυτές οι ελλείψεις πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι λοιπόν το δικό μας συμπέρασμα ότι ο τρέχον μηχανισμός συνεργασίας δεν επιτρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά τα θέματα αυτά. Η πρόταση της, νομικής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνεται και σε προηγούμενες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίως η το ψήφισμά σας του περσινού Μαρτίου για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Εσείς συστήσατε τότε, πρώτα, να εναρμονιστούν οι μηχανισμοί και μεθοδολογίες HTA, δεύτερον, να στοχευθούν σε θεραπευτικές πτυχές και να γίνουν υποχρεωτικέ οι σχετικέ αξιολογήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά ευθυγραμμίζονται πολύ με την ίδια την οτροπία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το λόγο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τι ειλικρινεί ευχαριστίε μου προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα προ τη δική σα Επιτροπή διότι η δική σα υποστήριξη υπήρξε πολύ σημαντική όλα τα τελευταία χρόνια και η συμβολή σα έχει μεγάλη αξία. Θα ήθελα τώρα να σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση του ουσιαστικού περιεχομένου της προτάσεως που βεβαίω θα συζητηθεί αργότερα με λεπτομέρεια. Οι συστάσεις σας έχουν αποτελέσει τη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στόχευση στις κλινικές πτυχές. Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία εκεί μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή κοινέοι μηχανισμοί και διαδικασίες HTA σε όλες τις χώρες μέλη. Να εργαστούμε δηλαδή από κοινού σε τέσσερις βασικούς τομείς. Πρώτα, κοινέ κλινικές αξιολογήσεις ε, ε, φαρμάκων και ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεύτερον, κοινέ επιστημονικές διαβουλεύσεις, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν αυτοί που αναπτύσσουν σχετικές θεραπείες, τεχνικές και ε, ιατρικές συσκευές, τι απαιτείται. Τρίτο, εντοπισμός των αναφιωμένων τεχνολογιών, αυτό που λένε στα αγγλικά horizon scanning, σάρωση του ορίζοντα για να βρούμε ποιε υπόσχονται να επιτύχουν. Και τέταρτο, η κυριοθέληση, η εθελοντική συνεργασία και πέραν του υποχρεωτικού εύρους φάσματος της ε, εφαρμογής της οδηγίας. Το βασικό χαρακτηριστικό της προτάσεώς μας είναι η δημιουργία ενός οργανωτικού νομικού πλαισίου για τις χώρες μέλη για να μπορούν να κάνουν κοινέ αξιολογήσεις νέων καινοτόμων τεχνολογιών σε σύγκριση με αυτές που ήδη υφίστανται. Οι κοινέ αξιολογήσεις θα γίνονται για φάρμακα τα οποία περνούν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αδειοδοτήσεων, ιδίως για νέες ενεργές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν για νέες θεραπείες. Για τις ιατρικές συσκευές το πεδίο εφαρμογής θα είναι περιορισμένο σε ορισμένα προϊόντα υψηλού κινδύνου όπου έχουμε λάβει ήδη τις γνωμοδοτήσεις από τους εμπειρογνώμονες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά από αυτό, τα συμβούλια HTA στις χώρες μέλη θα επιλέγουν ένα υποσύνολο των προϊόντων αυτών για να γίνει μια κοινή αξιολόγηση η οποία θα βασίζεται σε συμπεφωνημένα κριτήρια όπως την ε, ενδεχόμενη επίπτωση στην υγεία των ασθενών και σε συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά στοιχεία τη προτάσεω μα είναι να διασφαλίσουμε ώστε η συνεργασία ξεκινά από τι ίδιε τι χώρε μέλη, να εξασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα και έγκαιρη απόδοση των αξιολογήσεων, να χρησιμοποιούνται δηλαδή οι αξιολογήσει από τις χώρες μέλη στις δικές τους αξιολογήσεις, αλλά οι χώρες μέλη θα συνεχίσουν να διεξάγουν τις δικές τους εθνικές αξιολογήσεις των οικονομικών και άλλων μη κλινικών πτυχών, που είναι πιο συγκεκριμένες και σημαντικές για να βασίζονται εκεί οι εθνικές αποφάσεις. Οι χώρες, ε, μέλη, η HTA των χωρών μελών, θα λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού στην ομάδα συντονισμού. Κάθε χώρα μέλος θα εκπροσωπείται στην ομάδα αυτή και μάλιστα θα έχει ισότιμη ψήφο. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε με το όραμά μας, ότι η πρότασή μας δηλαδή είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τεχνολογιών του ιατρικού τομέα. Αυτό προβλέπεται και στη σταδιακή εφαρμογή που προβλέπει η πρόταση που θα επιτρέψει έτσι τις χώρες μέλη να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα. Θα έχουν τη δυνατότητα να ε, συμμετέχουν, να ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα και να συμβάλλουν με τις δυνάμεις τους στην κοινή προσπάθεια σε μια αύξηση της συνεκτικότητας των αξιολογήσεων. Και κάτι το οποίο θα αυξήσει και τη διαφάνεια με τη συμμετοχή και ενδιαφερομένων μερών όπως ε, ασθενών, κλινικών και ούτε καθεξής. Θα προαχθεί έτσι η επένδυση σε σχετικές τεχνολογίες, κάτι που θα είναι προστιθέμενη αξία υπέρ των ασθενών, θα αποδείξει τη δυνατότητα καινοτομία και αυτή θα αποβεί επίση υπέρ των ασθενών, διότι οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο της προτάσεως που έχει ως στόχο μια πιο αποτελεσματική και διαφανή αξιολόγηση των ιατρικών ή τεχνολογιών υγείας υπάρχει μεγάλο δυναμικό στην πρόταση για να διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες που θα επιτρέψουν στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις βέλτιστες δυνατές τεχνικές. Γνωρίζετε ότι τους τελευταίους δύο μήνες είχα μια σειρά διμερών συναντήσεων με πλήρωνες ευρωβουλευτές για να εξηγήσω τις προθέσεις της προτάσεως και για να ακούσω τις προκατακτικές τους απόψεις ορισμένων εξημών βασισμένη στις ανταλλαγές αυτές απόψεων και έχοντας απαντήσει σε πολλές από τις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να τονίσω τα εξής. Πρώτο, ναι, και η συμμετοχή και η επικαιροποίηση των κοινών αξιολογήσεων τεχνολογιών υγείας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά, ώστε να αποφευθεί οι χώρες μέλη να επαναλαμβάνουν τις κλινικές αξιολογήσεις σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερο, θα ήθελα επίσης να καθησυχάσω τις ανησυχίες σχετικά με τις ιατρικές συσκευές. Τονίζω ότι η πρότασή μας δεν έχει στόχο να επιβάλλει νέες απαιτήσει σε αυτούς που αναπτύσσουν νέες ιατρικές τεχνολογίες πέραν αυτών που υπάρχουν ήδη σε εθνικές νομοθεσίες. Βοηθούμε επίσης να αποφευθεί η αβεβαιότητα σχετικά με το πρόσθετο ενδεχόμενο γραφειοκρατικό βάρος Τέλος, η πρόταση θα λάβει υπόψη την αποκεντρωμένη πρόσβαση σε ε, θεραπείες και ε, ιατρικές συσκευές. Τέταρτο, το κόστος θα είναι περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Προϋπολογισμό όταν το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις χώρες μέλη, έχω συναντηθεί και με πολλούς υπουργούς υγείας για να τους εξηγήσω την πρόταση Πρόσφατα, επίσης, η Βουλγαρική Προεδρία έκανε μια πρώτη συνάντηση ομάδας εργασίας, όπου παρουσιάσαμε την πρότασή μας, η οποία έγινε ευμενώς δεκτή. Δυστυχώς, η Προεδρία προβλέπει μόνο δύο ακόμη συναντήσεις μέσα στους επόμενους μήνες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να οργανωθούν και άλλες τέτοιες συναντήσεις μέχρι το καλοκαίρι. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, απευθύνω έκκληση προ εσά να εμπλακείτε επικοδομητικά και να κάνετε, να υλοποιήσετε την πρωτοβουλία αυτή που θα αποβεί, όπως είπα, υπέρ των ασθενών. Ε, να ορίσει εισηγητή και συνεισηγητέ στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό για να αρχίσουν οι καρποφόρε συζητήσει μαζί μα. Υποστηρίζουμε και ε, μάλλον, ε, αναμένουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θέλουμε να δοθεί τελική μορφή στην νομοθεσία αυτή πριν από το 2019, δηλαδή την ημερομηνία των ευρωεκλογών. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να κάνουν τις ερωτήσεις τους και θα ξεκινήσω με τους ε, εισηγητές. Ο κύριος Λίζε πρώτος, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους, έχουμε την πρόταση. Την υποστηρίζω καταρχήν. Την περιμέναμε άλλωστε πολύ καιρό. Πραγματικά είναι σημαντικό να αποφευθεί η διπλή δουλειά, η επικάλυψη και για σας θα είναι καλύτερα και για τη βιομηχανία βεβαίως θα είναι καλό να αποφύγει τις επικαλύψεις αυτές. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, πώς μπορείτε να ορίσετε το όριο μεταξύ των καθηκόντων της κοινή αξιολόγησης HTA, τι θα γίνει δηλαδή από κοινού και τι θα παραμείνει στην αρμοδιότητα των χωρών μελών. Αυτό πρέπει να ε, διευκρινιστεί. Δεύτερη ερώτηση βρίσκω σημαντικό να μιλήσουμε όχι μόνο για το ερώτημα τι πράγμα θα αξιολογηθεί ακριβώς μετά την αδειοδότηση κλινικά, αλλά να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και των ε, αρχών HTA. Και βλέπω εδώ στο άρθρο 3 για επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Να Περιοριστούμε δηλαδή σε αυτά που πραγματικά έχουν μια προστιθέμενη αξία. Να γνωρίζει δηλαδή και η βιομηχανία τι αναμένει να πράξει. Τέλος, κάτι που δεν αναφέρεται σε αυτήν την πρόταση, γιατί και αυτή η πρόταση νομίζω δεν είναι επαρκή εν υπάρχει μια αξίωση που έχει επαναλάβει η παρούσα Επιτροπή, κίνητρα για ε, καινοτόμες δράσεις στον χώρο των αντιβιωτικών σιγά σιγά αρχίζω και ε, γίνομαι ανυπόμονος διότι όλοι λένε από τον πρόεδρο της Επιτροπής μέχρι και τα κατώτερα επίπεδα ότι το θέμα βιάζει. Ρωτώ λοιπόν τον Επίτροπο εάν μπορούμε ακόμη φέτος να αναμένουμε νομοθετική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χάνονται καθημερινά ανθρώπινες ζωές διότι δεν δραστηριοποιούμεθα έγκαιρα. Έχει έρθει η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Νταλή. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Αντριουκάητης που ήρθατε και μας παρουσιάσατε και αυτή την πρόταση. Ξέρετε και εσείς πως για μας το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η αξιολόγηση αυτής της τεχνολογίας θα αποτελέσει ένα κρίσιμο σημείο της κανονιστικής νομοθεσίας και για τα ιατρικά προϊόντα και για τις συσκευές και εμείς οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες εδώ και καιρό ζητάμε ε, μια τέτοια αξιολόγηση η οποία θα είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό μάλιστα το έχουμε τονίσει και στην πρόσφατη ε, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, πρόσβαση στα φάρμακα. Είμαστε πολύ σταθερή σε αυτά που ζητάμε εδώ και καιρό, γιατί με τον τρόπο αυτό, με αυτή την αξιολόγηση, θα μειωθούν οι ανισότητες, θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση η οποία σε επίπεδο κόστους θα είναι πολύ πιο ε, θετική, ε, μια και δεν θα κάνουν όλα τα κράτη-μέλη τις ίδιες αξιολογήσεις, τις ίδιες τεχνολογίες. Παρόλα αυτά, έχω κάποιες ερωτήσεις για τις οποίες θα ήθελα να μου απαντήσετε, γιατί ακόμα, για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποιο θα αναλάβει την αξιολόγηση. Είπατε πως έγιναν συζητήσεις για το θέμα και αναφερθήκατε σε κάποιες σκέψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τώρα, η Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Φαρμάκου δεν θα είναι υπεύθυνη. Για ποιο λόγο. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση και το χρονοδιάγραμμα. Επίσης με απασχολεί, ε, λάβαμε αργά στην διάρκεια αυτής της θητείας προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να πείτε πώς θα εξασφαλίσετε πως ως ε, διαιτητής ο οποίος διευκολύνει την όλη διαδικασία θα προσέξετε έτσι ώστε η διαδικασία να κυλήσει ομιλά, ομαλά για να διευκολύνουμε και να προχωρήσουμε με αυτή την νομοθεσία. Και έχω και μία τελευταία παρατήρηση είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να σας συνοδεύσουν σε αυτή τη διαδικασία. Είστε πεπισμένους πως θα ευεργαμιστούν τα κράτη-μέλη μετά όσα προτείνετε. Ε, είστε σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πιέρκα είναι ο επόμενος ε, ομιλητής από την ECR. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι πολύτιμη. Έχουμε καιρό που περιμέναμε τη σχετική πρόταση και για την αξιολόγηση της ε, τεχνολογίας αυτής όλα τα θέματα είναι σημαντικά. Συμφωνώ με τους στοχευμένους με τις στοχευμένες περιγραφές στο έγγραφο, συμφωνώ με τις λεπτομέρειες και στις λεπτομέρειες για την εναρμόνιση ε, πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε ε, με μεγάλη περιέργεια τα όσα θα επιλέξετε γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τις αλληλοπικαλύψεις μεταξύ κρατών μελών όταν πρόκειται για την ίδια φαρμακευτική τεχνολογία. Έτσι θα μειώσουμε το κόστος αλλά θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Είναι εξίσου σημαντικό οι επιστημονικές δυνατότητες και το τεχνολογικό δυναμικό ε, των διαφόρων περιφερειακών ε, υπηρεσιών να ε, ληφθούν υπόψη στο βαθμό που υπάρχουν, γιατί ξέρετε πως είναι διαφορετικά τα επίπεδα στις διαφορετικές περιοχές και η προσέγγιση που προτείνεται είναι να ομαδοποιηθούν σε ένα συμβουλευτικό, σε ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο και να προσπαθήσουν να καταλήγουν πάντα σε ένα κοινό συμπέρασμα. Δεν είναι κακή αυτή η πρόταση, αλλά προκύπτουν τα εξή θέματα. Καταρχήν, η επιλογή των ιατρικών τεχνολογιών που θα αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτές οι οποίες θα αξιολογούνται σε εθνικό επίπεδο. Πώς κάνετε ε, το διαχωρισμό. Γιατί εδώ, για παράδειγμα, έχουμε την χειρουργική τεχνολογία, η οποία είναι διαφορετική και εξίσου σημαντική. Όταν μιλάμε για ιατρικές συσκευές, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εδώ έχουμε μια τεράστια παραγωγική βάση, με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θεωρώ ότι αυτές που είναι πανευρωπαϊκές είναι λίγες. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει κάποια στοιχεία να μείνουν εκτός της ευρωπαϊκής αξιολόγησης γιατί έχουμε και ηθικές, ε, ηθικά προβλήματα και οικονομικά προβλήματα όταν ε, συζητάμε κάποιο είδους τεχνολογίας. Οπότε θα πρέπει να δίνεται και δυνατότητα εξαίρεσης. Επίσης, να δούμε η καινοτόμως τεχνολογία. Πώς θα επιλέγεται. Στηρίζω το γεγονός πως δεν θα εμπλακεί στην όλη ε, διαδικασία Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου γιατί περιμένω ε, και εγώ να δω πώς θα μοιραστούν οι αρμοδιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, πρόταση, λέει η κυρία Μάισνερ. Πρέπει να σας πω πως όσα μας περιγράψατε είναι πολύ λογικά. Είναι Καλή ιδέα να έχουμε αυτή την κοινή αξιολόγηση. Είναι πιο απλό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχω τις εξής τρεις ερωτήσεις. Τώρα, αντιθέτως από ότι για τα φάρμακα δεν υπάρχει κεντρική αδειοδότηση στην Ευρώπη. Το έχετε λάβει αυτό υπόψη στην πρότασή σας. Δεύτερο, διαφορετικές προϋποθέσεις, απαιτήσει των χωρών μελών για τις κλινικές μελέτες. Χρειάζεται λοιπόν, είναι, χρειάζεται λοιπόν μια δημοκρατική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με συμμετοχή των χωρών μελών. Πρόκειται για κεντρικό θέμα όμως, η μεθοδολογία δηλαδή των ιατρικών προτύπων. Δεν το βάζετε όμως αυτό στην ίδια την πρότασή σας, αλλά στα παρατήματα. Και τρίτη ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα της κεντρικής μεθοδολογίας με διαφορετικές όμως προϋποθέσεις αναχώρα μέλος. Ευχαριστώ κύριε Κονέτσουνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνατε κύριε Επίτροπε. Η πρότασή σας αποτελεί ένα βήμα προς την κατάλληλη κατεύθυνση Έχετε, χάρηκα που άκουσα ότι έχετε λάβει υπόψη τις προτάσεις του περσινού μας ψηφίσματος. Κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. Δεν συμβαίνει συχνά από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν συμβαίνει, ξαναλέω τόσο συχνά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις μας. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Όμως ταυτόχρονα δηλώνω ε, λίγο απογοητευμένη, διότι Μιλείτε για την υποχρεωτική αποτίμηση των, ε, του κόστους των ιατρικών προϊόντων. Θεωρώ όμως ότι από την αρχή υφίσταστε μεγάλη πίεση από τις παλιές χώρες μέλη, οι οποίες δεν θέλουν να μπει το στοιχείο, το στοιχείο του κόστους μέσα στην νομοθετική σας πρόταση. Όμως οι μικρές χώρες αυτό ακριβώς θα ήθελαν. Η δική μου χώρα, η Τσεχική Δημοκρατία, ε, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με τις τιμές των ιατρικών φαρμάκων. Όταν η χώρα μου διαπραγματεύεται τις τιμές ε, των φαρμάκων, δεν έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα γιατί είναι μικρή χώρα. Υπάρχει και το πρόβλημα εξάλλου των παραλλήλων επανεξαγωγών. Διότι εν τέλει άλλες χώρες πλουτίζουν από τα δικά μας συστήματα υγείας. Ελπίζω η πρόταση που έχετε καταθέσει δεν θα αποδυναμωθεί. Οι στόχοι που έχετε θέσει είναι και για μας σημαντικοί. Τι εννοώ. Θα πρέπει η νομοθετική πρόταση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας. Αυτό είναι σημαντικό. Ελπίζω το ίδιο να αντιληφθεί η Βουλγαρική Προεδρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συμβάλλει. Ελπίζω θα μας υποστηρίξετε και εσείς και ότι και οι χώρες μέλη θα καταβάλουν την αναγκαία προσπάθεια ώστε η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους της κοινοβουλευτικής θητείας. Διότι τότε θα έχουν και οι χώρες μέλη επαρκή χρόνο για να δράσουν και ελπίζω ότι τότε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για το γεγονός που μας παρουσιάσατε αυτό το σχέδιο εδώ. Δεν θέλω να σας κρύψω πως η σημασία του θέματος είναι τέτοια γιατί έχουμε τη συναχή ε, μεταλλαγή της τεχνολογίας της ιατρικής και της φαρμακευτικής που αναμένουμε ε, μου δημιουργεί πάρα πολλούς προβληματισμούς και η ίδια η μεθοδολογία σας επίσης γιατί έχουμε μεν τις ιατρικές συσκευές ε, που πρέπει να αξιολογήσουμε, αλλά έχουμε και τις τεχνικές που ακολουθούν οι ιατροί, οι νοσηλευτές και νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε τι γίνεται ε, με την αναγνώριση των ε, ιατρικών διπλωμάτων και βέβαια το γεγονός ότι έχουμε αυτή την αναδυόμενη τεχνολογία ε, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί δεν γνωρίζουμε καθόλου ποιες θα είναι οι εξελίξεις τα επόμενα 5-10 χρόνια και οι επιπτώσεις για τους ασθενείς είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε σφαιρικά. Δηλαδή η σχέση μεταξύ νοσηλευτή, ιατρού και ασθενή θα αλλάξουν πάρα πολύ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Και βέβαια εσείς μιλήσατε για τη διάσταση την νοσοκομιακή, την κλινική, ε, την ιατρική, υπάρχει όμως και η ηθική. Οπότε, αν έχουμε αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ που θα ε, δαπανούμε κάθε χρόνο, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως θα πρέπει ε, οι ασθενείς να δρέψουν τα πλεονεκτήμα αυτής της αξιολόγησης και όχι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και οι, τα εργαστήρια τα οποία μέσω της τεχνολογίας και της ρομποτικής και τα λοιπά θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Νομίζω πως θα πρέπει εδώ να εξασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως τα ιατρικά πτυχία θα είναι τα ίδια σε όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνει έτσι ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τον Επίτροπο για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Και μετά θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Να ξεκινήσω από τον Πίτερ Λίζε και την ερώτησή του. Πώς μπορούμε να χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ κλινικών και μη κλινικών θεμάτων. Κατά την άποψή μου είναι σαφής η πρόταση και καταδεικνύει σαφέστατα ότι ακολουθούμε την αρχή της επικουρικότητας διότι όταν αναφερόμαστε στις ε, δυνατότητες ε, να συζητήσουμε την, τα θέματα τιμολόγησης και αποζημίωσης, αυτό επαφίεται στα κράτη-μέλη. Ε, και επίσης, θέματα αναλογικότητας. Η πρότασή μας είναι ιδιαίτερα αναλογική και δεν θέλει να παρέμβει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αλλά η πρότασή μας βασίζεται στον κανονισμό της εσωτερικής αγοράς Και αν το εξετάσουμε από το πρίσμα της εσωτερικής αγοράς, ακολουθούμε το άρθρο 114 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ αντιλαμβανόμαστε σαφέστατα τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών και προτείνουμε μόνο εθελοντική συνεργασία εάν κάποιες χώρες αποφασίσουν ότι ε, δεν μπορούν να κάνουν πλήρη ε, αξιολόγηση τεχνολογίας ε, βάσει κλινικού και μη κλινικού πεδίου, μπορούν να την κάνουν από κοινού με άλλες χώρες, ιδίως στους τομείς των πολύ σπάνιων ασθενειών, όπου δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ασθεν... αριθμός ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί μπορεί κανείς να ε, δει ότι μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να γίνει μια οικονομική αξιολόγηση έχοντας μια πλήρη εικόνα. Και η πρότασή μας βασίζεται σε αυτό. Η υποχρεωτική συμμετοχή ε, υπάρχει μόνο στον τομέα των κλινικών ε, δοκιμών, ε, στον τομέα των μη κλινικών δοκιμών, εκεί επαφείται στα κράτη-μέλη και αυτό μας επιτρέπει να προτείνουμε και μια ρήτρα διασφάλισης, ε, διότι κάποιες χώρες έχουν τις ιδιωτερότητές τους και μπορούν να κάνουν επαναξιολόγηση της κλινικής αξιολόγησης, αλλά θα πρέπει αυτό να είναι δεόντως αιτιολογημένο, να το κοινοποιήσουν και από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν συγκεκριμένα κριτήρια και να κάνουν επιπλέον κλινική αξιολόγηση εφόσον θεωρούν ότι συντρέχει λόγος. πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτούς που αναπτύσσουν φάρμακα και ιατρικά προϊόντα να διαθέσουν κονδύλια για νέες τεχνολογίες. Η πρότασή μας εξετάζει ε, το ενδεχόμενο καταρχάς να υπάρχει το λεγόμενο horizon scanning και επίσης να δοθούν κάποιες δυνατότητες ε, να έρθουμε σε επαφή και διαβούλευση με αυτούς που αναπτύσσουν τα φάρμακα και να τους κατευθύνουμε και να τους δώσουμε συμβουλές ε, κατά τον επενδυτικό του σχεδιασμό για να δούμε ε, ποιες ε, νέες τεχνολογίες είναι στον νοδρίο ζωντά ή στα σκαριά. για τα αντιβιωτικά και νέους μηχανισμούς για κίνητρα για έρευνα για τα αντιβιωτικά. δεν είμαι ακόμα σε θέση να απαντήσω αυτή την ερώτηση, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει την έκθεση για την αναθεώρηση όλων των μηχανισμών που παρέχουν κίνητρα στη διάθεσή μας. Θα περατωθεί όμως στο τέλος του έτους και θα εξετάσουμε και τις δυνατότητες για μια κοινή εικόνα και κάποιες νέες πρωτοβουλίες. Έχω μιλήσει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τις δυνατότητες να αναπτύξουμε ε, ε, νέες έρευνες, ε, να έχουμε κάποιους νέους επιστήμονες και νέους ανθρώπους που αναπτύσσουν φάρμακα που να ασχολούνται με τα θέματα και να εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να οργανώσουμε ίσως και μια στρογγυλή τράπεζα το φθινόπορο, για να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά ε, να αντιληφθούμε πώς έχει κατάσταση μεταξύ των διαφόρων μοντέλων για κίνητρα και να έχουμε και κατά νου και διάφορες δυνατότητες για να υπάρχει μια καθοδήγηση για τα νέα μοντέλα ε, για κίνητρα. Περιμένουμε όμως τα τελικά αποτελέσματα της έκθεσής μας που θα μας δώσει και κάποιες ε, κατευθύνσεις. Ερωτήσεις της κυρίας Ντάλη τώρα. Γιατί δεν ελήφθη υπόψη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαραμάκων, ο EMA. Πρέπει να πω ότι έχουμε μια γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην δημιουργήσουμε νέα προσκόμματα για την υγεία. Υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι είχαν, ήταν κατά της συμμετοχής ε, του οργανισμού φαρμάκων στις ε, νέες τεχνολογίες για την υγεία. Η ιδέα μας είναι να ε, συγκροτηθεί μια μόνιμη γραμματεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επειδή ε, η διαδικασία αυτή μπλέκει και τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να μας παρουσιάσουν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν ποια τεχνολογία θα πρέπει να αξιολογηθεί και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία από πολύ νωρίς. Ένας κοινό μηχανισμός επιστημονικής διαβούλευσης. Ο οργανισμός φαρμάκων θα συνεργαστεί ε, με αυτούς τους φορείς ε, αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, αλλά τα πρώτα στάδια της ε, διαδικασίας της ε, κεντρικής ε, έγκρισης για τα φάρμακα ε, θα βασίζονται στην ίδια αρχή ε, στην οποία βασίζονται και σήμερα, όπως προβλέπετε σήμερα με τους διάφορους φορείς ε, για την τεχνολογία για την υγεία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Όσον αφορά το πόσο έγκαιρα θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, έχετε δίκιο, πρέπει να προτρέψουμε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν δυνατότητες και να μας τις παρουσιάσουν για να ολοκληρωθεί η πρόταση πριν από τις ευρωεκλογέ. Και σας διαβεβαιώ ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Έγιναν και συζητήσεις πριν ε, καταρτήσουμε την πρόταση και τώρα έχουμε συζητήσεις ε, και προτρέπουμε τα κράτη-μέλη για να καταλάβουν και ποιος είναι ο στόχος μας ε, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρόταση. Διότι στην όλη διαδικασία έχουμε μια εξαετία. Τρία χρόνια για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιτροπολογίας και από εκεί και πέρα τρία χρόνια για να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ε, στο νέο τρόπο συνεργασίας. Βεβαίω πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να διαβουλευτεί με τα κράτη-μέλη, να διευκολύνει τη διαδικασία και να είναι ο εγγυητής πολύ καρποφόρων συζητήσεων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη, να τα ενημερώνουμε και να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις και να συζητούμε τα θέματα σε τεχνικό επίπεδο. Επίσης, τέτοια ερώτηση πώς μπορούμε να επιλέξουμε τις νέες τεχνολογίες. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια διαδικασία της οποίας ηγούνται τα κράτη-μέλη. Από τη μια προτείνουμε να συσταθεί αυτή η ομάδα η οποία θα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει ε, πώς έχει η κατάσταση παντού, ε, να κάνει το horizon scanning. Αυτοί από εκεί και πέρα θα παρουσιάζουν στη συντονιστική ομάδα τι μέλη γενέστε, τι τεχνολογίες ε, θα προκύψουν στην επόμενη τριετία, πενταετία ή δεκαετία. Και από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν ποιες τεχνολογίες θέλουν και θα επιλέξουν να τις ε, συμπεριλάβουν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας τους και στη συνέχεια αυτό θα επιτρέψει και στη συντονιστική ομάδα να ξεκινήσει αυτές τις κοινέ ε, κλινικές αξιολογήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία επιλογής είναι στα, είναι στα χέρια των κρατών μελών. Αλλά βεβαίως η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων είναι απαραίτητη, διότι η διαδικασία έγκρισης για τη διάθεση στην αγορά είναι κεντρική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο μόνος τρόπος να συνεργαστούμε με τη Συντονιστική Ομάδα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων είναι αυτός και προτείνεται σαφέστατα στην νομοθετική μας πρόταση. Η κυρία Μάισνερ έθεσε κάποιες ερωτήσεις για ε, ευρία δημόσια συζήτηση και δυνατότητα να εγγυηθούμε δημοκρατική διαφάνεια. Ναι. Ε, θεωρούμε ότι στην όλη διαδικασία των τεχνολογιών υγείας μπορούν να συμμετέχουν οργανώσεις ασθενών, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, γιατί πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση για τα κλινικά πρότυπα, τις προδιαγραφές και τη δυνατότητα να δούμε ποια ε, κλινικά στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Η δυνατότητα επίσης να συμπεριλάβουμε ε, κάποια κριτήρια που αφορούν την προστασία των δεδομένων των ασθενών. Ε, και φυσικά ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να παρέχουν πληροφορίες και να συνεργαστούν στον τομέα των κλινικών δεδομένων και θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα. πάντα με γνώμονα τι νέε απαιτήσει ε, για την προστασία δεδομένων. Σίγουρα βέβαια χρειάζονται συζητήσεις ε, δημοσίως από αυτό και είμαι βέβαιος ότι οι οργανώσεις ε, ασθενών και τα πανεπιστήμια μπορούν να συμβάλλουν στον τομέα αυτό και να είναι και ιδιαίτερα δραστήριοι. Η κυρία να έθεσε κάποιες ερωτήσεις για το πώς μπορούμε να έχουμε ε, πλήρη αξιολόγηση της τεχνολογίας για την υγεία. Συμφωνώ μαζί σας ότι σε κάποιους τομείς ε, σπάνιων ασθενών, όταν έχουμε πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό ασθενιών, ασθενών συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, συντρέχει λόγος να γίνει μια οικονομική αξιολόγηση. Για παράδειγμα, στην Κύπρο ή στη Λιθουανία, όταν έχουμε 100 άτομα οι 300 άτομα, 300 μόνο ασθενείς που πάσχουν από κάποια συγκεκριμένη νόσο ε, και γνωρίζουμε ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 18.000. Σίγουρα πρέπει να γίνει μια πανευρωπαϊκή οικονομική αξιολόγηση ε, και κοινωνική αξιολόγηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό μας βοηθά να έχουμε μια οικονομία κλίμακας ε, σε συζητήσεις με τον κλάδο για την τιμολόγηση αλλά πρέπει να δείτε και το θέμα της εθελοντικής συνεργασίας στον τομέα αυτό. Προτείνεται αυτή η προαιρετική συνεργασία ε, στην οποία τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν ε, να ε, κάνουν κάτι από κοινού για τον εξή απλό λόγο ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφή οικονομική αξιολόγηση. ετέθηκε μια ερώτηση για την αναλογία μεγάλων ε, πολυεθνικών ε, επιχειρήσεων αφενός ε, και τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας και τη διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να εγγυηθούμε διαφάνεια και έτσι θα αυξήσουμε και την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπεία και δεν έχει σημασία από ποια ε, εταιρεία θα προέρθει η προτινόμενη θεραπεία. Ε, θεωρώ ότι η πρότασή μας μπορεί να μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ασθενών, να λαμβάνουν καινοτόμες θεραπείες και να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας τους και φυσικά να έχουμε σαφείς κανόνες και διαφάνεια στις συζητήσεις με τον κλάδο για ε, την τιμολόγηση και τις αποζημιώσεις. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε μόνο χρόνο για τέσσερις ερωτήσεις. Ελπίζω να μιλήσει για ένα λεπτό καθένας η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνοντας τη διαδικασία αξιολόγησης, μπορούμε να φανταστούμε πως θα επιταχύνουμε και την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτομίες της ιατρικής τεχνολογίας. Άρα λοιπόν είμαι σαφέστατα υπέρ. Σε κάποια κράτη-μέλη αξιολογήσεις σε μερικό βαθμό ε, χρηματοδοτούνται από κάποια τέλη. Τι θα γίνει λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Και βέβαια είναι και οι εθνικές, ε, εθνικοί φορείς αξιολόγηση που ανησυχούν για την ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από αυτή την ε, ε, χρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, γιατί δεν επιλέξαμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε κοινά προγράμματα εργασίας μεταξύ κρατών μελών. Επίσης, θεωρώ πως είναι πολύ ασαφής η διάκριση μεταξύ των ε, νοσοκομιακών δοκιμών και των οικονομικών στοιχείων τη στιγμή της αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας και θα ήθελα να πείτε αυτό το κομμάτι πώς θα το λύσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι γρήγορη κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που είναι πολύ σημαντική για όλους και για τα συστήματα εθνικής υγείας και νομίζω ότι ε, η βιωσιμότητα των συστημάτων μας βασίζεται στην ε, βελτίωση της έρευνας και της τεχνολογίας στην ιατρική. Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι λείπουν οι λεπτομέρειες από την πρότασή σας και από το έγγραφο ε, του οποίου θα εργαστούμε. Και νομίζω ότι για τις κλινικές αξιολογήσεις νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε στην τρέχουσα θητεία. Οπότε μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία θα πρέπει να μας επιτρέψει να είμαστε επιτυχείς. Άρα λοιπόν ποια είναι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα βελτιώσουμε την έρευνα και θα επιτρέψουμε πετύχουμε την απόλυτα απόλυτη πρόσβαση όλων των ασθενών ε, σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Γιατί δεν θα πρέπει αυτή η αξιολόγηση να πιέζει τα κράτη-μέλη να αδειοδοτήσουν μεν κάποιο φάρμακο, αλλά δεν εξασφαλίζει παράλληλα πρόσβαση σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαντίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, είχα κάποια άλλα πράγματα και παρακολουθούσα από το γραφείο μου. Χαίρομαι και εγώ για αυτή την ε, πρωτοβουλία, διότι ε, πιστέψαμε σε αυτήν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ξέρω πώς σκοπεύει ο Επίτροπος να πείσει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία. Διότι εμείς θέλουμε κάτι το οποίο να είναι αποτελεσματικό, επομένως υποχρεωτικό διότι ακούγονται ε, κάποιες χώρες που έχουν ιδιαίτερους δισταγμούς. Πάντα υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με τα κράτη-μέλη που διστάζουν ε, να δεχτούν ε, κάποιες προτάσεις. Ε, πιστεύετε ότι ε, ένα πλήρες ε, τεχνολογικό σύστημα υγείας που περιλαμβάνει και ε, συγκεκριμένα προφίλ θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη για συγκεκριμένα φάρμακα. Έχω κατά νου τα ορφανά φάρμακα σε αυτή την περίπτωση. Η κυρία Κάντεμπαχ. Πρώτα σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και εμείς ε, χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την πρόταση της Επιτροπής. Εξ αρχής θα άλλαζα ωστόσο τον τίτλο της να κάνετε αντί CHTA, δηλαδή πρόκειται για την κλινική αξιολόγηση των ε, τεχνολογιών υγείας. Κλινική αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, διότι γενική μπορεί να γίνει μόνο εάν ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις. Δεύτερο, όπως λέχθηκε και από άλλους προηγουμένως, υπάρχει ένα σύνολο ρυθμίσεων για το πώς γίνεται ή λαμβάνονται οι αποφάσεις στις διάφορες αυτές ε, ε, ομάδες συμβούλων, εμπειρογνωμόνων κλπ. Υπάρχουν ε, γίνονται ψηφοφορίες. Και τέλος, εκεί όπου υπάρχουν ή προβλέπονται δεσμευτικά καθήκοντα, θα υπάρχουν μακροπρόθεσμα και κυρώσεις. Θα προβλέπονται και κυρώσεις. Προβλέπεται μηχανισμός επιβολής κυρώσεων εάν οι χώρες δεν ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το γύρο ερωτήσεων. Ε, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Θα ξεκινήσουμε την ερώτηση κυρίας Κάτεμπαχ για τον ορισμό λείπτουμε και τα δύο. Δηλαδή και το κλινικό και το μη κλινικό και εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να κάνουν πλήρη αξιολόγηση προσφέροντας και εναλλακτικές ε, δυνατότητες μέσω συνεργασιών. Προσωπικά πιστεύω ότι για, κάποια, για κάποιους πολύ μικρές οι σπάνιες παθήσεις να έχουμε το, την πλήρη αξιολόγηση. Για παράδειγμα, όταν είπα ότι μπορεί να υπάρχουν 17.000 μόνο ασθενείς ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε γιατί να το κάνουμε ξεχωριστά την οικονομική αξιολόγηση σε κάθε ένα κράτος μέλος διαφορετικά. Αλλά θα πρέπει να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν το σκέλος αυτό, γιατί βέβαια Υπάρχουν κοινωνικοί, οικονομικοί, οργανωτικοί, νομικοί, ηθικοί λόγοι που διαφέρουν μεταξύ μας. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως υπάρχει μια ευκαιρία να ξεπεραστούν αυτές οι διαφορές και να παρουσιάζουμε ε, κοινή, πλήρη τεχνολογική αξιολόγηση. Συμφωνώ μαζί σας. Πάντως αυτό που προτείνουμε τώρα είναι μόνο αυτή την πολύ ρεαλιστική προσέγγιση ακριβώς γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη αντίσταση σε διάφορους χάρους. Μία ψήφος αναχώρα είναι η απάντηση στην άλλη ερώτηση, οπότε αν υπάρχει συνένεση σίγουρα το καλύτερο, αλλά και απλή πλειοψηφία. Διαφορετικά χρησιμοποιείται ειδική πλειοψηφία με μικρές μειοψηφίες που μπλοκάρουν οπότε θα αποφασίσει ο συνομοθέτης ή συνομοθέτης αλλά για μας απλή πλειοψηφία συνένεση ή απλή ψηφία. Κυρία Καβεσόν, για τις περισσότερες λεπτομέρειες που ζητήσατε, συμφωνώ μαζί σας και σε κάποιες περιπτώσεις όντως χρειάζονται, αλλά ας κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων και ειδικά σε θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα, γιατί ξέρετε πως καμιά φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ποιο είναι το όριο μεταξύ ε, του νοσοκομιακού και μη νοσοκομιακού. Οπότε ας το κάνουμε μεταξύ μέσω εφαρμοστικών και κατεξουσιδότηση πράξεων, να τα συζητήσουμε σε τεχνικό επίπεδο και αν προτείνετε εσείς κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, συμφωνώ έτσι ώστε να ενισχύσουμε ε, τη σαφήνεια αυτής της πρότασης. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε πραγματικά να βελτιώσουμε τα, ε, τη σαφήνεια αυτής της πρότασης. Κυρία Γκαρτίνη, πώς θα πείσουμε τα κράτη-μέλη Ένα εργαλείο έχω μόνο. Στα χέρια μου και αυτό είναι η υπομονή. Η υπομονή και οι ασθενείς. Γιατί τελικά οι ασθενείς είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν πρόσβαση σε θεραπείες. Είναι τα δικαιώματα των ασθενών. Of course, all Και θα πρέπει να το κατανοήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί όλη η προσπάθειά μας βασίζεται στο ότι υπάρχουν ασθενείς. Και θα πρέπει να τους δοθεί πρόσβαση σε καινοτόμοι, καινοτόμες θεραπείες, γιατί πολλές φορές η πραγματική ε, η πραγματικότητα πια είναι ότι από την έγκριση μέχρι τη θεραπεία μπορεί να περάσουν και 7 και 5 χρόνια, οπότε ναι, υπάρχει το θέμα της πρόσβασης των ασθενών. Πρέπει τα θέματα αυτά να τα συζητήσουμε. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαστε εδώ ακριβώς προς όφελος των ασθενών. Και βέβαια γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως κάποια κράτη έχουν τα δικά τους εθνικά συστήματα και πολλά επιχειρήματα, αλλά ευθυγραμμαζόμαστε εδώ με τα εθνικά του συστήματα και κυρίως για τις μεγαλύτερες χώρες έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία να ε, εκπροσωπήσουμε τα, όλα τα κράτη-μέλη ανεξάρτητα με το που βρίσκονται οι ασθενείς, σε μικρά κράτη-μέλη, σε μεγαλύτερα. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να παροτρύνουμε το Συμβούλιο να δράσει και βασίζομαι στην Βουλγαρία για να γίνουν περισσότερες συναντήσεις κατά την Προεδρία της πριν δώσει τη σκητάλη στην Αυστρία. Ξέρω πως η Αυστρία πραγματικά ενδιαφέρεται για το θέμα και είμαι αισιόδοξο. Ε, για το κατά πόσο θα μπορέσουμε να πιέσουμε και να πείσουμε τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε αποτελέσματα. Και για την τελευταία ερώτηση, ναι. Για τα τέλη τα οποία θα μπορούσαμε μετά να μοιράσουμε σε εθνικό επίπεδο, ναι. Βέβαια, δεν μπορούμε εμείς να προτείνουμε κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να έχουμε μια ειδική ε, επιδότηση που θα πληρώνεται στη χώρα γνωμοδότη, για παράδειγμα, μέσω του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού. Μας ρωτήσατε γιατί δεν επιλέξαμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ξέρετε πως πολλά κρατημέλη έχουν εδώ διαφορετικές απόψεις και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ειδική πλειοψηφία που θα μας επιτρέψει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οι προτάσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες και φορείς και οργανισμούς αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται από όλους εμάς να δούμε ποιες είναι οι καινούριες προτάσεις, τι συμπεριλαμβάνουν Πάντως πρέπει να σας πω πως είμαι πολύ προσεκτικός πριν προτείνω κάτι καινούριο. Ευχαριστώ πολύ. και για τη διαθεσιμότητά σας και για το ότι πιέσετε όλες τις ε, ερωτήσεις. Είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε όλα αυτά με καινούριες ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ. we can Να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε τις ε, κάρτες σας για την ψηφοφορία. Αν είστε έτοιμοι, η πρώτη ψηφοφορία είναι για την ένσταση ή αντίρρηση για συστήματα εχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού του κυρίου Μαρζή. Θα γίνει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία η οποία αρχίζει τώρα. Τέλος. Απορρίπτεται, όπως βλέπετε. Δεύτερο, ένσταση σχετικά με την διάθεση στην αγορά γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού με διάφορους αριθμούς. Ενία ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Κάποιος ε, παρατηρεί από την αίθουσα ότι δεν πρόλαβε να βάλει την κάρτα του. Ένσταση σχετικά με την ανανέωση εγκρίσεως για τροποποιημένο καλαμπόκι με άλλους αριθμούς. ενία ψηφοφορία αρχίζεται. Πέρας. Μία ψήφος περισσεύει των φιλελευθέρων, των Άλντε. Καλώς τώρα. Εγκρίνεται η εν λόγω ένσταση. ψηφοφορία για την ε, συνολική απαγόρευση χρήσης πειραματοζώων για καλλιντικά. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ή επαλήθευση επαλήθευση για την 22 αρχίζει πέρας εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 τμήμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ε, συγγνώμη απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ 56 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται αυτή 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει Πέρας και εγκρίνεται. Πολύ καλά. Η επόμενη τώρα που είναι και η τελευταία. Ψηφίζουμε την πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου του Νιουκάσλ. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά επίσης αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί η εντολή. Όχι. Καλώς. Ωραία λοιπόν. Αυτά. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Θα σας δω σήμερα το απόγευμα. Και καλή σας όρεξη.